Συνεχίζουμε με την Αιθιοπία ε, πλέον σε ανοιχτή συνεδρίαση. Η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας ε, επέκρινε την Αιθιοπία σε πολλά σημεία για περιορισμού στην κοινωνία των πολιτών, μαζικές συλλήψεις, ε, διαδηλωτών και δημοσιογράφων, καθώς επίσης και μελών της αντιπολίτευσης. Επίσης έκανε λόγο ε, για εκτελέσεις ε, χωρίς δίκη. Το τέλος του 2015 η Αιθιοπία αντιμετωπίζει ένα κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ε, που κλιμακώθηκαν από τις αρχές του 2016 και μετά σε διάφορες ε, ε, πόλεις και περιοχές της χώρας και διαδηλώσεις οι οποίες διαλύθηκαν με τη βία σε πολλές περιπτώσεις από τις αρχές. Στις αρχές Οκτωβρίου δεκάδες ίσως και εκατοντάδες άτομα έχασαν την ζωή τους σε μια μαζική φυγή ε, ατόμων ε, κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στην Αντισαμπέμπα ε, από ό,τι φαίνεται η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει δακρυγόνα και πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης και αυτό προκάλεσε τα, το θάνατο αυτών των ανθρώπων. η κυβέρνηση κήρυξε κατάκτηση έκτακτης ανάγκης όλη τη χώρα για έξι μήνες σήμερα καλέσαμε εμπειρογνώμονες, ειδικού για θέματα της Αιθιοπίας, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέλιξ Χόρν. Ε, είναι ε, ειδικευμένο ερευνητής ε, για θέματα του ΚΟΝ της Αφρικής για την Human Rights Watch. Παρακαλώ. Thank you for this opportunity to speak. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε μια κρίσιμη στιγμή στο Κοινοβούλιο και κρίσιμη και για τους δυο μας. Στις 2 του Οκτώβρη, άγνωστος αριθμός ατόμων, πιθανώς εκατοντάδες, πέθαναν μετά από τη χρήση δακρυγόνων, από τις δυνάμεις ασφαλείας στα πλαίσια ενός φεστιβάλ μιας θρησκευτικής γιορτής που περιλαμβάνει εκατομμύρια προσκυνητές. Αυτό οδήγησε σε οργή σε όλη την περιοχή της Ορομίας. Υπήρξαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και καταστροφή κυβερνητικών κτηρίων και ιδιωτική περιουσίας αυτών που θεωρείται ότι ήταν κοντά στο καθεστώς. Στις 9 του Οκτώβρη ο Πρωθυπουργό κήρυξε μια κατάσταση εκτάσεις ανάγκης εξάμεινη και τα πρόσφατα συμβάντα Ακολούθησαν 11 μήνες διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης, κυβέρνηση η οποία είχε προτείνει ένα νέο ρυθμιστικό για την Αντίσα Βέμπαν, κάτι το οποίο έπλητε τους γεωργούς, κάτι το οποίο γινόταν ε, και τα περασμένα χρόνια και σε άλλα μέσα εθεπιείας. Ολόκληρη λοιπόν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ακύρωση αυτού του ρυθμιστικού και υπήρξε δίκη της ανταπόκρισης των δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις. Όπως επίσης και υπήρξαν καταγγελίες ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής του Ορομόξ. Είχαμε πολλές οικογένειε και συγγενείς οι οποίοι συνελήφθησαν ή εξαφανίστηκαν. Τον Ιούλιο είχαμε μεγάλες ε, διαδηλώσεις και σε άλλες περιοχές λόγω εθνοτικών χαρακτηριστικών και είχαμε και πάλι συγκρούσεις με αυτούς που είχαν σχέση με το κυβερνών κόμμα. Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 100 άτομα σε ένα αιματηρό Σαββατοκύριακο. Τώρα, όπως προχωράνε τα συμβάντα, οι εξελίξεις, οι... μπορέσαμε να εντοπίσουμε το πώς χρησιμοποίησαν υπερβολική και θανατηφόρο βία οι δυνάμεις ασφαλείας σκοτώντα 500 ε, ανθρώπους και πολλοί χιλιάδες ε, κρατήθηκαν χωρίς να κατηγορία. Είχαμε λοιπόν ευρεία χρήση βασανιστήριων και δολοφονιών μέσω στρατιωτικών δυνάμεων στις οποίες ανατέθηκε η επαναφορά της τάξης μετά από αυτά τα συμβάντα. Η Αιθιοπία λοιπόν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες κρίσεις της από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, ανέλαβαν καθήκοντα κυβερνήσεις το 1991. Το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι αντικείμενο πίεση προς την κυβέρνηση όσον αφορά τις παραβιάσεις και εμεί θα πρέπει να δώσουμε ανάλογα. Τα πρόσφατα συμβάντα δεν έγιναν ξαφνικά. Είχαν οριμάσει. Ήταν το αποτέλεσμα της κυβερνητικής υπολογισμένης συστηματικής παραβίασης βασικών ελευθεριών και καταπίεσης της, του δικαιώματος έκφρασης και των ελευθεριών. Είχαμε φυλάκιση ε, δημοσιογράφων, bloggers και δημοσιογράφων οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ σύλληψη. Ε, ή άλλων ε, κυρώσεων. Πολύ συχνά δεν τους επιτρέπεται να κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί που παρέχουν πληροφορίες στους ξένους δημοσιογράφους συλλαμβάνονται. Τους τελευταίους τρεις μήνες μπλόκαρε το ίντερνετ πλήρως η κυβέρνηση. Περιόρισε την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και σταμάτησε τις ε, εκπομπές συμπαραβομένης και της Deutsche Welle. Έχουμε αναφορές ε, περιορισμού της πρόσβασης στην χώρα όσον αφορά την ηλεκτρονική πρόσβαση μετά από αυτό που έγιναν. Ομάδες από την, από την κοινωνία των πολιτών αντιμετωπίζουν παρόμοια αντιμετώπιση. Είχαμε ήδη συμβάντα τα οποία περιόρισαν την δυνατότητα δράση των ΜΚΟ. Είχαμε ένα νόμο κατά της θερμοκρατία το 2009 που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης ε, ακτιβιστών, δημοσιογράφων και άλλων οι οποίοι ε, καταδικάστηκαν χωρίς δίκη και φυλακίστηκαν. Είχαμε επίσης σοβαρού σοβαρούς περιορισμούς στην δράση των πολιτικών κομμάτων, κάτι το οποίο ε, επέτρεψε στην τονίση συμμαχία να κερδίσει τις εκλογές του Μάη 2015 με 100% των ψήφων παρά βεβαίως ε, τις ε, αντικυβερνητικές έτσι, διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. Και σε κάποιες, στις πιο εκλογές είχαμε το 99% και στις να με το 9%. Είχαμε επίσης συλλήψεις αυτών που ήταν πραγματικοί υποτιθέμενοι διοργανωτές των ταραχών και των διαμαρτυριών θεωρώ ότι υπάρχει και έχει επικρατήσει ο, ο φόβος. Διαδηλωτές, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους και χρησιμοποιήθηκε βία από τις δυνάμεις ασφαλείας πολύ συχνά. Όποιος δηλαδή αφισβητεί την κυβέρνηση ή διαμαρτύρεται ή είναι αντιφρονούντας ε, έχει συνέπειες η κυβερνητική πλειοψηφία καταπίεσε οποιαδήποτε αντίθετη φωνή. Συνελήφθη πρόσφατα ένας συνάδελφος μαζί με άλλους έξι όταν πήγαινε σε ένα κατάστημα τροφίμων στον Ναϊρόμπι και άλλοι συνάδελφοι, συνάδελφοι του κατηγορήθηκαν ότι ανήκαν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και ένοπλες οργανώσεις. Είχαμε και έναν μεταφραστή που δούλευε για την Παγκόσμια, Πράεδρα, σε ένα, ε, Παγκόσμια Τράπεζα σε ένα πρόγραμμα σε κάποια χωριά, το οποίο και αυτός ε, συνελήφθη. Είχαμε επίσης και τις υποχρεωτικές μετατοπίσεις ηθαγενών και χιλιάδες άτομα τα οποία έφυγαν από την Αιθιοπία και διέφυγαν στις ε, γειτονικές χώρες. Μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας χρηματοδοτείται αυτό το πρόγραμμα και, την Ένωση, και από την Ένωση και από άλλους η περίπτωση αυτού του μεταφραστή ήταν κλασική για όσους προσπαθούν να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση. Δηλαδή είχαμε συλλήψεις, βασανισμούς, άσκηση βίας, απλά και μόνο επειδή εξέφρασαν διαφορετική γνώμη. Αυτό αφορά όλους δασκάλους, ε, δημόσιους υπαλλήλους, όλους. Επίσης, καταγράψαμε και την τη χρήση της ε, αναπτυξιακή βοήθειας εκ μέρου τη κυβέρνηση της Αιθιοπίας όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων και τη βοήθειας ε, σε πρόσβαση ας πούμε στα φυτοφάρμακα, ε, απασχόληση, θέσει εργασία. Από το 2010 βλέπουμε ότι δεν έχει λάβει ιδιαίτερη δράση η Ένωση για την εποπτεία ακριβώς της κατάληξης αυτής της αναπτυξιακής βοήθειας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινομένα και σήμερα. Η αναπτυξιακή βοήθεια λοιπόν είναι πολύ χρήσιμη όσον αφορά την εξάλληψη της φτώχειας στην Αιθιοπία και σε άλλα μέρη. Αλλά βεβαίω υπάρχει αυτή η παρενέργεια, δηλαδή τη αυθαίρετης χρήση από την κυβέρνηση για να καταστήλει την ε, αντιπολίτευση. Και βεβαίως η κυβέρνηση αρνείται να τα συζητήσει όλα αυτά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έτσι μια ήρεμη διπλωματία στην ε, Αιθιοπία γιατί έχει ε, επιδεινωθεί η κατάσταση και είχαμε πολλές παραβιάσεις. Το να παραβλέψουμε την καταστολή της κυβέρνησης ε, σημαίνει ότι θα θέσουμε τις εταιρικές μας σχέσεις σε κίνδυνο όσον αφορά και θέματα όπως η μετανάστευση. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρξαν κάποια σημαντικά βήματα. Παραδείγματο χάνει το Γενάρη, το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα εδώ και χρόνια για το Κοινοβούλιο ζητώντα μια μετατόπιση τη πολιτική τη Ένωση, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν έχει συμβεί. Γι' αυτό ακριβώ ζητάμε από εσά σήμερα, σε στενή συνεργασία με του ομολόγου σα στα Εθνικά Κοινοβούλια, να πιέσετε την Ένωση και όσε χώρες γίνεται, ώστε να λάβουν ισχυρή και έντονη δράση για να μην επιδενθεί η κρίση στην Ευθυοπία. Η πρόσφατη ανακήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης νομίζω θα πρέπει να αναστραφεί. Υπό το Εθνές Δικαίο οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε μέτρα αφορούν την ε, ελευθερία έκφρασης και του εσωτερίζεσθε θα πρέπει να εξετάσονται και θα πρέπει να είναι ανάλογα με τους στόχους που επικαλείται η κυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να έχουμε καταπίεση δικαιωμάτων ή στιγματισμό ανθρώπων λόγω εθνότητας ή παραβίαση δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ζητήσουμε να μην χρησιμοποιείται βία και αυτή ακριβώς η κυβέρνηση, η ομή καταστολή όλων των αντιφρονόντων οδήγησε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Αιθιοπία. Υπάρχουν τρει κρίσιμε δράσει που πρέπει να λάβει η Ένωση βραχυπρόθεσμα. Καταρχά, θα πρέπει να συνεχίσει την διεθνή έρευνά τη όσον αφορά τα συμβάντα σε αυτές τις τρεις περιοχές ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 και τα πρόσφατα συμβάντα στο, στο θρησκευτικό, στη θρησκευτική γιορτή. Ήδη έγινε ένα πρωτοβήμα το Σεπτέμβριο θετικό, αλλά θα πρέπει η Ένωση να πιέσει την, Αιθιοπία, την να καλέσει διεθνείς επιθεωρητές και ερευνητές για να αποτιμήσουν τα συμβάντα αυτά. Η από το 2007 η Αιθιοπία δεν έχει ειδικού εισηγητέ ε, από τον ΟΗΕ, ενώ αντίθετα αυτό ισχύει με την Ερυθρέα. Δεύτερον, η Ένωση θα πρέπει δημόσια να ζητήσει από την Αιθιοπία να απελευθερώσει όλους αυτούς που κρατήθηκαν παράνομα. Και συγκεκριμένα είχαμε ένα άτομο το οποίο ήταν ε, εξέχον στέλεχος της αντιπολίτευσης και το οποίο ε, φυλακίστηκε επειδή ακριβώς εξέφρασε την αντίθεσή του στις, στις πολιτικές της κυβέρνησης και μάλιστα κατηγορήθηκε για τρομοκρατική δράση. Δεν θα πρέπει λοιπόν οποιαδήποτε δράση της Φρόντων να θεωρείται ως τρομοκρατική δράση. Επίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να άρει τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, όπως πρόσβαση στο ίντερνετ και παραμποδισμό των ε, δημόσιων μεταδόσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω ξανά το λόγο στην υπηρεσία εξωτερική δράση ε, και στην κυρία Κλάουντα, Κλάουντια Βίντε. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση του Φέλξ Χόρν. Έχουμε διαβάσει τις εκθέσεις της Human Rights Watch και της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς επίσης και άλλων διεθνών οργανισμών και οργανώσεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία. Συμφωνούμε ότι προκαλούν βαθιές ανησυχίες Έχουμε συζητήσει και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε να συζητάμε την κατάσταση με τους Αιθιοπές συνομιλητές μας εδώ στην Αντισαβέμπα και ε, οποιαδήποτε στα περιθώρια οποιασδήποτε διεθνούς ε, συνάντησης στην οποία βρισκόμαστε και ε, προσπαθούμε να δούμε και τις αιτίες και τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας ε, προσπαθεί να αναλύσει την κατάσταση και να εντοπίσει τις ε, αιτίες. Το, το πόρισμα, το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων εν μέρη έγινε γνωστό ε, σε τοποθετήσει του Προέδρου αλλά και στο Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι Σαφές όμως είναι ότι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί ως τώρα για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα ε, των ε, πολιτών δεν είναι επαρκής. Οι πολίτες δεν θεωρούν ότι οι ανησυχίες τους ε, εισακούστησαν. Οπότε, παρόλη την, παρόλο τον προβληματισμό της κυβέρνησης, παρόλα τα μηνύματα που έχει στείλει οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται και μάλιστα διευρύνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ε, βλέπουμε μια κλιμάκωση της βίας. Εσείς αναφέρατε τα δραματικά γεγονότα της ε, θρησκευτικής γιορτής ε, η Ρίτσα, όπου έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι αλλά εκτός από αυτό έχουμε δει και επιθέσεις ε, εναντίον ιδιωτικών επενδύσεων, ε, τουριστικών καταλημάτων. Πολλά από αυτά είναι χρηματοδοτούμενα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν χρηματοδοθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα προσφέρουν θέσεις εργασίας και απασχόληση. Όλα αυτά αποτελούν μια μαζική εκδήλωση απογοήτευσης ε, του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων. Όλοι γνωρίζουμε πως η κυβέρνηση αποφάσισε την ε, κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη αντιδράσαμε με μια δήλωσή μας, ζητήσαμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Επίσης ζητήσαμε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με τον λαό, με τους πολίτες και όχι απλώς να περνάει μηνύματα. Ζητήσαμε ο διάλογος να είναι ειλικρινής ε, και να ακουστούν οι ανησυχίε των πολιτών. Δημερός ε, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επαφή με αξιωματούχους των, της Αιθιοπίας και στις Βρυξέλλες και αλλού. Και ε, έχουμε εκφράσει την άποψή μας. Ε, ρητά. και έχουμε ζητήσει πράξεις έτσι ώστε να φανεί ε, το αν η αιθιοπική κυβέρνηση πραγματικά έχει προσήλωση στην ε, βελτίωση των, της επαφής με τον ε, λαό. Επίσης έχουμε προβλέψει έναν διάλογο σε υψηλό επίπεδο προκειμένου να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα, ιδιαίτερα την εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιούμε όποια ευκαιρία μας δίνεται για να οικοδομήσουμε έναν πραγματικό διάλογο με ανταλλαγή απόψεων, με δυνατότητα να κινητοποιήσουμε, να οθήσουμε και να ενθαρρύνουμε δράσεις σύμφωνες με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιστεύουμε ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί ή τα προβλήματα να λυθούν με τη χρήση βίας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάμε πάντα. Βέβαια εξετάζουμε το πώς θα επηρεαστούν οι διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιθιοπίας. Ε, μετά την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν είχαμε ακόμα το χρόνο να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα. Γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, αυτές οι επαφές. Είναι σαφές ότι όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις στις σχέσεις μας με την Αιθιοπία. Να πω και δύο λόγια για την ε, συμφωνία στρατηγικής δέσμευσης που υπογράφηκε με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, νωρίτερα το 2016. Αυτό αποτελεί ένα πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο για να εμβαθύνουμε τον διάλογο σε συγκεκριμένου τομεί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διακυβέρνηση είναι ένας από αυτούς του τομεί. Προ το παρόν δεν έχουμε ξεκινήσει την εφαρμογή της ε, συμφωνίας αυτής. Ε, πολλές ε, φορές είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση από τα λόγια, από τα κείμενα στις πράξεις. Ένας, μία δράση ήταν η διοργάνωση ενός φόρουμ επιχειρηματιών που είχε προβλεφθεί για τον Νοέμβριο. Τώρα αναβλήθηκε Είναι προφανώ, προφανώς ε, ακατάλληλη η στιγμή για να διοργανωθεί ένα, μια τέτοια εκδήλωση ε, μελλοντικών επενδυτών, ενδυνάμει επενδυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αιθιοπία. Ε, το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο. Οπότε στην πράξη δεν έχουμε ξεκινήσει καμία άλλη πτυχή της συμφωνίας στρατηγικής δέσμευσης. Όμως αυτή η συμφωνία είναι εργαλείο και έχουμε συμφωνήσει με την Αιθιοπία ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι η πρώτη από τις πτυχές που θα ξεκινήσουν ε, στην Αιθιοπία και ελπίζω ότι θα έχουμε και υψηλό επίπεδο παρουσία από τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πρέπει να στα τελειώσουμε στις 10.30 και έχουμε ακόμα και άλλους ομιλητές. Ο Hans Stausbol, καταρχήν, ε, τμήματάρχης στον συντονισμό ε, της ανάπτυξης Αφρική, της Ανατολικής Αφρικής. Ε, παρακαλώ πολύ σύντομα, διότι πρέπει να πάρουν το λόγο και η κυρία Μακάβαν και οι, ευρωβουλευτές. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και νομίζω ότι η Κλάουντι Συνάδελφο έχει δικαλύψει τα περισσότερα σημεία. Όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, ε, λειτουργούμε παράλληλα με το πολιτικό σύστημα, που, το πολιτικό πρόγραμμα που υπάρχει από την ΕΕΣ. Στα αναπτυξιακά προγράμματα ε, και με, αυτούς τους, με τις στρατηγικές ε, δεσμεύσεις προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο μας και θέλω να αναφέρω ότι η συνεργασία αφήνεται ε, βασίζεται στην εταιρική σχέση. Αυτή είναι η βασική αρχή και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Μαζί με την κυρία της Αιθιοπία καταφέραμε να υποστηρίξουμε μια διαδικασία που επέφερε πολλά ωφέλη στην ανάπτυξη για τους ανθρώπους της Αιθιοπία. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα προβλήματα, αλλά αν το συγκρίνουμε την κατάσταση του 83 και το 84, σε αυτή την περίπτωση δεν χρειαστήκαμε με τον πόνο για να έχουμε την κατάλληλη ανταπόκριση. Δεν χρειαστήκαμε έναν στάρ. Γιατί η κυβέρνηση της Αιθιοπίας καταφέρει να έχει κάποιες πρόοδους στην αναπτυξιακή πτυχή όσον αφορά τις κατηγορίες και τα λοιπά, γνωρίζουμε πολύ καλά την ησυχία που εκφράστηκε και υπάρχουν ε, μαρτυρίες σχετικές. Δεν ήταν ότι σταματήσαμε, την, ε, τη στήριξή μας εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Επίσης, θέλω να επιστήσω την προσοχή ότι παρόλο που συνεργόμαστε ε, στενά με την κυβέρνηση της ΕΘΠΕΣ, όλα τα προγράμματα ε, όλα τα προγράμματά μας ε, στοχεύουν αποκλειστικά στη βελτίωση της ζωή των πολιτών της Αιθιοπίας. Είναι οι κυρίως δικαιούχοι του καινούριου ε, ταμείου. 97 ε, εκατομμύρια θα πάνε στην Αιθιοπία και αυτά τα κονδύλια στοχεύουν την βοήθεια που θα παραχθεί σε άτομα που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη, όπως είναι οι πρόσφυγες που επηρεάζονται από την ξηρασία και από τις ε, συνθήκες ε, του εκτοπισμού γενικότερα, τις επιπτώσεις του εκτοπισμού. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, έχει εθνικό πρόγραμμα έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα 745 εκατομμυρίων ε, ευρώ Μέχρι στιγμή έχουν επιστοθεί τα 500 εκατομμύρια και θα προχωρήσουμε με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο προβλέπεται στο προγραμματικό έγγραφο που περιέχει συγκεκριμένε χρηματοπιστωτικέ διατάξει για την υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών. Καταλαβαίνω αυτό που είπε ο Φίλιξ. Ότι ναι, συνεργαζόμαστε εντό ενό πλαισίου που περιορίζει τι δυνατότητέ μα δεν το αρνούμαστε, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε και πιστεύω ότι υπάρχει κατανόηση από την πλευρά τη κυβέρνηση να ε, ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Θα σταματήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο για λίγα λεπτά στην κυρία Μπέτρη Μιέσου, υπεύθυνη για το κράτο Αφρική από την Γενική Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Θα αναφέρω, όπως γνωρίζετε, ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είμαστε μερόληπτοι και ουδέτεροι και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε συγκροσμένοι με την κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε με ανθρωπιστική κρίση εδώ, που δεν μπορεί φυσικά να κατονομαστεί ακριβώ έτσι σε ανθρωπιστική κρίση, όμω ε, επί τη ουσία περί αυτού πρόκειται. Όσον αφορά την ασφάλεια που σχετίζεται με το Ελληνίνιο, ναι, σίγουρα ε, δεν ήταν επίπεδο Ελληνίνιο αυτό που έγινε. Δεν είναι πω πριν από 10-15 χρόνια. Όμως και το 2015 και το 2016 ήταν σημαντικές επιπτώσεις. 17 ε, εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από αυτό, 1,5 εκατομμύρια χρειάστηκαν ανθρωπιστική βοήθεια. Υπήρξε πρόγραμμα κυβερνητικό για την παροχή βοήθειας. Δεν αναφέρθηκαν ε, οι εντός της χώρας εκτοπισμένοι πληθυσμοί πάνω από 700.000 εκτοπισμένοι λόγω διαφόρων αιτιών, αιτιών για θέματα επιστηστικής ασφάλειας κτλ. Και φυσικά αυτό αναφέρθηκε, είναι η προσφυγική κρίση. Η Αιθιοπία είναι η μεγαλύτερη χώρα φιλοξενίας προσφύγων. 741.000 πρόσφυγες έχει περίπου είναι από την Νότια, ε, Νότιο Σουδάν, από την Ερυθρέα, από τη Σομαλία. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να πω η υπόθεση της Ερυθρέας. Δεν μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για πρόσφυγες που προσπαθούν να διαφύγουν από μια δύσκολη κατάσταση, μια σύραξη στη χώρα της και που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους αν μεταστραφεί η κατάσταση. Δεν είμαστε αφελείς και πρέπει να παραμείνουμε ουδέτεροι, ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι. Όμως παράλληλα παρακολουθούμε στενά όχι τόσο πολύ τις συγκρούσεις που δεν επηρεάζουν το δικό μας πρόγραμμα, αλλά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ανάλογα με τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε σε διάφορες περιοχές όπου έχουμε προγράμματα, εκπονούμε προγράμματα για να δούμε ποια είναι η πρόσβαση των ανθρωπιστικών εταίρων και για να έχουμε αυτή την πρόσβαση πρέπει, πρέπει να έχουμε την πρόσβαση, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε την εξολόγηση, να κάνουμε την παρακολούθηση των προγραμμάτων και γι' αυτό χρειαζόμαστε άμεση πρόσβαση στις περιοχές αυτές γιατί διαφορετικά πρέπει να σταματήσουμε τα προγράμματα και το δεύτερο είναι η ασφάλεια. Δεν έχουμε αποδεικμένο αντίκτυπο ε, στους ε, εταίρους μας, αλλά αν υπάρξει πρόβλημα τους δικούς μας ε, εταίρους, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην Αιθιοπία. Αυτός ο χρόνος είναι ένας ιδιαίτερος χρόνος από την πλευρά, από την πλευρά της χρηματοδότησης, γιατί ε, έχει γίνει πίστοση μεγαλύτερο ποσού για την Αιθιοπία από ό,τι σε προηγούμενα έτη. Δίνω το λόγο τώρα στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, κυρία Μακάβαν. Ε, είμαστε πολύ πιασμένοι από το χρόνο, θα είμαι πολύ σύντομη. Η, Γενική Διεύθυνση ε, Ψηφιακής Βοήθειας ε, μας είπε ότι η Αιθιοπία είναι ε, η χώρα στην οποία πηγαίνουν τα μεγαλύτερα κονδύλια αναπτυξιακής βοήθειας. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνει ιδιαίτερε προσπάθειες να είναι σταθερή χώρα και να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες. Όλοι οι πολιτικοί γνωρίζουν πως αντιπολίτευση υπάρχει πάντα. Ακόμα και μέσα στο ίδιο σου το κόμμα πολλές φορές έχεις ε, αντιπολίτευση. Αυτό αποτελεί τμήμα της ζωής, είναι κάτι το φυσιολογικό, θα πρέπει να το δέχονται όλοι. Γνωρίζω το Ελνίνιο, γνωρίζουμε την δύσκολη κατάσταση στην Αιθιοπία, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, όμως ε, δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε θα πρέπει η αντιπολίτευση να αναγνωριστεί ως ε, μια ε, πραγματικότητα και θα πρέπει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα της αντιπολίτευσης με τρόπο δημοκρατικό, ε, ειρηνικό και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό θα περάσει στους Αιθιοπές και ελπίζω θα, μπορούμε να, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια δημοκρατική σταθερή Αιθιοπία που θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση της ευημερίας του λαού της. Ευχαριστώ. Δύο άτομα έχουν στήσει το λόγο. Κυρία Γκόμης, κυρία Λόχ Μπίρερ. Από ένα λεπτό. Θα τα καταφέρετε νομίζω. Θα... Ήθελα πράγματι να πιστέψω την αφελής η Κομισιόν, γιατί αλλιώς αν δεν είναι αφελής είναι ψεύτες η κατάσταση στην Αιθιοπία είναι τόσο άσχημη όσο την περιέγραψε ο κ. Χόρν. Δεν είναι δημοκρατική χώρα. Μόνο το, εθνικό, πρόσωπος του εθνικού μετόπου που ήταν εδώ ε, αντιμετωπίζει την Αιθιοπία ως νέα δημοκρατία. Είναι μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση ε, δεν έχει δημοκρατική νομοποίηση, δεν εξελέγει και σκοτώνει τον κόσμο. Είναι ντροπιαστικέ οι δηλώσεις αυτές, όπως αυτή που έχω στα χέρια μου. Πιστεύετε πράγματι ότι το Κοινοβούλιο είναι χώρος διαλόγου, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ε, δεν πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ο κ. Φέλξ Χόρν Μα ε, μας μίλησε για τις συστάσεις της Human Rights Watch είναι εξαιρετικές. Θα πρέπει να ζητήσουμε να γίνει ανεξάρτητη διερεύνηση των επεισοδίων, να ζητήσουμε την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων και των περιορισμών του ίντερνετ και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς επίσης να ζητήσουμε και την απελευθέρωση των φυλακισμένων μεταξύ αυτών και μελών της αντιπολίτευσης και άλλες συλλήψεις έγιναν και χτες αφότου επέστρεψε η κυρία Μέρκελ από εκεί και μας ντρόπιασε όλους μαζί. Κυρία Λοκπίλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν είναι δυνατόν θέλω να θέσω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο του Human Rights Watch. Μας είπατε για την κατάσταση, τον όρομος. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τους Σουγκαντίν. Και το δεύτερο ερώτημα αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει... δεν είναι επικαιρή πλέον. Ξεπερνάει την πραγματικότητα. Δεν κατονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνετε λόγο για το ταξίδι της κυρίας Μέρκελ επισκέφθηκε ε, ε, ε, συνάφθηκε μια συμφωνία με πέντε χώρες που δέχονται πρόσφυγες. Τις τρεις τις έχει, έχει επισκεφθεί. Ήδη η κυρία Μέρκελ. Όμως το παρασκήνιο είναι ότι δεν ασκούμε κριτική στην Αιθιοπία για, και στις άλλες χώρες για να κρατήσουν τους πρόσφυγες στο έδαφος τους. Και έτσι η σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές επηρεάζεται. Αν όμως δεν αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση την παραφύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα έχουμε προβλήματα και θέματα. Και θα επανερχόμαστε σε αυτά τα θέματα συνεχώ εδώ στην Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. κυρία Δεξιά και μετά ο κ. Αντάκτησον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με την ε, και την Βάρβαρα Λόχπιλερ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χόρν για την παρουσίαση που μας έκανε. Και ανησυχώ και εγώ για τα αποτελέσματα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Εσείς ε, μας αναφέρατε την κατάσταση πριν την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε καταλαβαίνουμε πώς θα είναι τώρα. Αντιλαμβάνομαι τις απόψεις της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, και των εκπροσώπων της Κομισιόν, αλλά υπάρχουν και όρια. λένε ότι οι αφρικανικές χώρες δεν καταλαβαίνουν την αιμονή μας, την αιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, δεδομένης κατάστασης εκεί βέβαια αυτό το καταλαβαίνουμε. Ε, οι μετακινήσεις των πληθυσμών είναι τεράστιες ε, και καταλαβαίνω, καταλαβαίνουμε γιατί δεν κατανοούν την άποψή μας. Ε, όταν έχουμε εκλογές που δίνουν σχεδόν 100% των ψήφων σε ένα κόμμα, καταλαβαίνει κανείς τι άλλο να πούμε. Αυτό δεν θα έπρεπε να μας χτυπήσει κόδωνα κινδύνου και να μας οδηγήσει στο να αλλάξουμε λίγο τη στάση μας. Με, το, με σεβασμό βέβαια. Υπό την προπόθεση όμως ότι δεν γελιο, γελιοποιούμαθα. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση γελιοποιείται αυτή τη στιγμή. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ούτε ψεύτες ούτε αφελείς, είναι κοινικοί απλώς οι συνομιλητές μας. Από όλα αυτά που μας είπατε κύριε Χόρν, αυτό που μου έμεινε είναι το θέμα της ιχνηλασιμότητας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Αιθιοπία, γιατί παίζεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίζεται η αξιοπιστία και των επιτόπιων συνομιλητών μας. Οπότε εκεί πρέπει να δουλέψουμε και χαίρομαι για το ζευγάρι σε εισαγωγικά που προεδρεύει τη συνεδρίασή μα, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάκτισον, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα αλλά σας περάσω να μιλήσω και σουηδικά. Ε, για αυτά που είπαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαμε ένα πολύ γνωστό Σουηδό γιατρό που πριν τρία χρόνια συνελήφθη στην Αιθιοπία με την κατηγορία ότι είχε συμμετάσχει σε κάποιες έτσι δράσεις διαφθοράς. Κατηγορήθηκε για διαφθορά λοιπόν. Η Σουηδική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι αθώος και ότι οι κατηγορίες που του απεγγείλαν ήταν πολύ ύποπτες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την εξωτερική δράση. Γνωρίζει αυτή την υπόθεση δεν μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, να κάνουμε κάτι αυτό το Σουηδό γιατρό. Bueno, tengo un gravísimo. Κοιτάξτε, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα χρόνου και θορύβου. Όσοι είστε λοιπόν εδώ στην αίθουσα, παρακαλώ κάνετε ησυχία. Η διπλωματική αντιπροσωπεία της Αιθιοπίας ζήτησε το λόγο για δύο λεπτά λόγω κοινοβουλευτικής αγροφροσύνης θα δώσουμε αυτό το χρόνο ομιλίας στις διπλωματικές αποστολές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε να το κάνουμε γραπτό στην προηγούμενη συνάδελφα. Θα δώσω δύο το λόγο, ε, για δύο λεπτά το λόγο στην ε, διπλωματική αντιπροσωπεία της Αιθιοπίας. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου Καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον και την ανησυχία της για την τωρινή κατάσταση στη χώρα μου. Να αποφεληθώ της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και την Ένωση για την συνεχή υποστήριξη, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Όπως ξέρετε, είναι η Ένωση ένας από τους κύριους εταίρους ανάπτυξης Συνεργαζόμαστε σε τομείς όπως κλιματική αλλαγή, μετανάστευση κλπ. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε πραγματικά αυτά τα πρόσφατα συμβάντα με τις ταραχές, αλλά ξέρουμε όλοι ότι όλες αυτές οι ταραχές χειραγωγήθηκαν από αντιφρονούντα στοιχεία που ζουν στην Ευρώπη και, την, και τη ΣΥΠΑ. Είχαμε απολύες ζωών, καταστροφή περιουσιών και έλλειψη ασφάλειας για τους πολίτες μας. Η χώρα μας εκφράζει την λύπη της για την απώλεια ζωών και τις καταστροφές. Και κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρούμε ότι η άσκηση του δικαιώματος δημοκρατίας της, ε, ε, στην Αιθιοπία δεν είναι κατά το δοκούν. Θα πρέπει να προσπίζουμε κυρίως τη χώρα και τους πολίτες μας. Από τη στιγμή που υπήρξαν ταραχές δεν είχαμε άλλη λύση από το να ασκήσουμε την δημοκρατία πλήρως και πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε ως μια χώρα με μια φωνή ενιαία. Θεωρούμε, Πρόεδρε, ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε δημοκρατία. Πιστεύουμε στον διάλογο πιστεύουμε στις συζητήσεις, στις επαφές. Όπως είπε και η Κλάντια προηγουμένως, θα το κάνουμε αυτό. Όμως δεν πιστεύουμε στην εισαγωγή δημοκρατίας. Ο λαός θα πρέπει να το αποφασίζει και θα πρέπει να αποφασίζει για το πώς θα ασκήσει η δημοκρατία του. Πριν 25 χρόνια ξεκινήσαμε την εφαρμογή της δημοκρατίας στην χώρα μας και τα 25 χρόνια αυτά πετύχαμε θετικά αποτελέσματα στον τομέα τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε πολλέ ε, εθνικέ και περιφερειακέ εκλογέ και οι μειονότητε εκπροσωπούνται με ρετούς στα κλακμένα μα σώματα. Έχουμε επίση έχουμε επίσης θεσπίσει και ένα δύο μεσολαβητή. Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει κάνει θαυμάσια δουλειά με έρευνε μετά από συστάσει των οργανισμών. Έχουμε αναπτύξει και ένα σχέδιο δράση και το έχουμε εφαρμόσει ανάλογα. Βεβαίως συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις, αλλά θεωρούμε ότι σε συζήτηση με την ομάδα σας θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δώστε μου μισό λεπτό ακόμα για να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Φέλεξ προηγουμένως σε σχέση με τις ε, διακρίσεις των κατοίκων της περιοχής Ορομός. Αυτοδικείται αυτή η περιοχή του Ορομός. Στο κοινοβούλιο εκπροσωπούνται οι κάτι με, σε ποστό 32%. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι από αυτή την εθνότητα. Έχουμε και υπουργού από την περιοχή του Ορομός, οπότε δεν καταλαβαίνω για ποια διάκριση μιλάτε. Και τέλος, σε σχέση με την εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Να σας διαβεβαιώσω ότι η λειτουργία της ανθρωπιστικής βοήθειας εφαρμόζεται σωστά στην Αιθιοπία και έχει διασφαλιστεί η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και η ελευθερία των ε, πολιτών σε συνεργασία βέβαια με τους υπουργούς και την κυβέρνησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην Αιθιοπία. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ του συναδέλφου που συμμετείχαν σε αυτή την κοινή ακρόση και θα συνεχίσουμε την ε, ημέρα.